Ja, liebe Kolleginnen συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, auf, uh, θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στο εκλεγέν Κοινοβούλιο. Συγχαίρω όλους τους συναδέλφους που εκλέγονται, επανεκλέγονται ή εκλέγονται για πρώτη φορά ε, ε, και θα Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για την καλή μας συνεργασία ε, τα τελευταία δυόμιση χρόνια πριν πω στην ουσία. Νομίζω στον έλεγχο του προπολογισμού πραγματικά καταφέραμε να κινήσουμε κάποιες καταστάσεις. Ε, ε, ο έλεγχος του προπολογισμού είναι δημοκρατικός έλεγχος των κονδυλίων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι κάναμε καλή χρήση αυτού του ελέγχου. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εκείνους που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί τους τα τελευταία δυόμιση έτη. Λοιπόν, ερχόμαστε στην εκλογή αυτή καθ' αυτή του νέου προεδρίου, του νέου προέδρου της νέας προέδρου της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να εκλέξουμε το Προεδρείο της Επιτροπής. Πρώτα θα εκλέξουμε τον Πρόεδρο ή την Πρόεδρο και τέσσερις στη συνέχεια την Πρόεδρος σύμφωνα με τον κανονισμό μας και το άρθρο 204. Θα πρέπει πρώτα να ελέγξουμε πόσοι δικαιούνται να ψηφίσουν. Νομίζω η γραμματεία μπορεί να μας πει ε, και για ποιους αναπληρωτές έχουμε ενώπιον μας που θα ψηφίσουν. Αν δεν απατώμε είναι δύο αναπληρωματικά μέλη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Δύο αναπληρωτέ από το ΕΛΚΑ έχουμε, έτσι δεν είναι. Ξέρουμε και τα ονόματα. Ο κύριος Φαντακάμπ και Πιτέρα, ο κύριος Πιτέρα. Α, ο κύριος Πίπερ, όχι Πι, τι γράφεται εδώ. Sorry. Okay, it's okay. Mm Okay. Um, in Group. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Τρεις αγνοούνται. Έχουμε τρεις αναπληρωτές παρόντες. Ποιοι είναι οι αναπληρωτές των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Παρακαλώ, κυρία Γιώτοβα έχει το λόγο. Α, είναι αναπληρώτρια μάλλον, κυρία Γιώτοβα. Yeah. Mr. Mr. okay. Ο κύριος Καταλίν. Και ο συνάδελφος Νίτερ Μούλερ παρόν. Ωραία. Οι λοιπές ομάδες, ΙΣΙΑΝ. Ο κύριος Κιόλβεν, αναπληρωτής. Ο κύριος Τσαρνέσκι, παρίσταται. Και ποιον αντικαθιστά τον κύριο Μπράτμπορν, μάλιστα. Φιλελεύθεροι, όλοι παρόντες. Γκουε, ο κύριος Ιόγκ. Η κυρία Κάρη απουσιάζει. Πρασίνους έχω δει και ο κύριος Σόλτες. Η FDD, Άνοτ. Okay. And, uh, Madame... Και η κυρία Μπεγκέν. Μία εγγεγραμμένη. Ο Λουί Αλιό. Μάλιστα. Ωραία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Παρακαλώ ε, τις υποψηφιότητες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, λέει ο κύριος Σάρβαμα, προτείνω την κυρία Ίγκιμπορκ Γκρέσλε, υποψήφια για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν? Όχι. Μπορούμε να ψηφίσουμε διαβοής λοιπόν. Εάν συμφωνείτε και δεν υπάρχουν αντίθετες ψήφοι. Συγχαρητήρια κυρία Γκρέσλε. Εκλέγεστε πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και ευτυχή θητεία και παρακαλώ να έρθεις να αναλάβεις την Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την απόδειξη εμπιστοσύνης. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και τον Μίχαηλ Τόιρερ και για το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο ήμιση της θητείας που ήταν ε, εξαιρετικό στην Προεδρία ε, και αυτό ε, βελτίωσε πάρα πολύ και τη φήμη μας στο Κοινοβούλιο. Και αυτό ε, σε δικαιώνει και για κάποιες δυσκολίες που γνώρισε και χαίρομαι που παραμένει μέλος στην Επιτροπή μας. Περνούμε στη συνέχεια στην εκλογή των αντιπροέδρων. Έχουμε προτάσεις για υποψηφίους. Έτσι, η τάξη πάνω απ' όλα. Και μάλιστα η Ισπανίδα το είπε αυτό το πράγμα. Έχουμε προτάσεις για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Sí, eh, bueno, en κυρία Γκρέσλερ. Ο δικός μας υποψήφιος για την πρώτη αντιπροεδρία της Επιτροπής είναι ο κύριος Ντέρεκ Βόν. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες προτάσεις. Όχι. Επειδή δεν έχει ζητήσει κανείς μυστική ψηφοφορία, ε, κύριε Ίσο, εκλεγέντε τον κύριο Βότ και τον συγχαίρω ε, ε, για την εκλογή του και χαίρομαι για τη συνεργασία που θα έχουμε. Πάμε στο δεύτερο αντιπρόεδρο. Έχουμε προτάσεις υποψηφιότητες. Ο Μπαρτ Στάζ, ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Προτείνω για δεύτερο αντιπρόεδρο το νέο συνάδελφο Ίγκορ Σόλτες, η του δεύτερου αντιπρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες προτάσεις έχουμε? Όχι. Και πάλι επειδή ζητεί κανεί μυστική ψηφοφορία, διαβοή εκλέγεται ο κύριος Σόλτες. Παρακαλώ ελάτε στο Προεδρείο και χαιρόμαστε για τη συνεργασία που θα έχουμε. Zum Για τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου, ο κύριος Τόιρερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευράς φιλελευθέρων προτείνω τη Μαρτίνα Γκλαμπάιωβα. Ευχαριστώ. Άλλες προτάσεις? Όχι. Και πάλι δεν έχει ζητηθεί μυστική ψηφοφορία, οπότε διαβοής ε, κλέγεται η κυρία Γλαμπάιοβα. Τέταρτος αντιπρόεδρος. Eh, Για τη θέση του τέταρτου αντιπρόεδρου προτείνουμε τον κύριο Νταν Νίκα, οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Μάλιστα, άλλη πρόταση υπάρχει. Όχι. Και πάλι δεν έχει ζητηθεί μυστική ψηφοφορία, οπότε μπορούμε διαφορείς να εκλέξουμε τον κύριο Νίκα. Συγχαρητήρια. Ελάτε παρακαλώ και εσείς στο πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι και προσβλέπω στη συνεργασία με όλους σας και με τα εκλεγέντα μέλη του Προεδρείου. Έχουμε βασική δουλειά μας εδώ την απαλλαγή για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε φορά. Αυτή η δουλειά είναι ακόμα μπροστά μας, επίκειται. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να σας ενθαρρύνω είναι πολύ σημαντική αυτή η δουλειά για τους φορολογούμενους μας και θα πρέπει και πολύ επιθετικά και πολύ συνειδητά να ε, τα παρακολουθείτε αυτά τα θέματα. Οι παλιοί τα γνωρίζουν. Για τους νέους θέλω να πω ότι οι φορολογούμενοι μας ε, χρειάζονται τη δική σας ε, στράτευση σε αυτό το σημείο και στην Επιτροπή μας. Πάμε στο σημείο 3. Προσεχή συνεδρίαση την 3 22 Ιουλίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30 το απόγευμα. Υποθέτω ότι η γραμματεία θα σας στείλει ένα πακέτο ε, καλωσορίσματος, αυτό το welcome package που βγάζουμε, για να γνωρίζετε τα πρώτα βήματα στην Επιτροπή μας. Δεν ξέρω αν έχετε καν μια παρατήρηση, πρόταση, κριτική να εκφράσετε, όχι. Τότε να κηρύξω το πέρα συνεδρίασης και πάλι χαίρομαι για τη συνεργασία μας και προβλέπω σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ.